Και ε, τώρα προχωρούμε στην μέσα διάταξη. Έχουμε το τελικό σχέδιο της μέσα διάταξη που σύμφωνα με το άρθρο 149 ε, έχει διανεμηθεί όπως για τη διάσκεψη των Προέδρων και επίσης έχουν ζητήσει τα κρατημέλη τι οι πολιτικέ ομάδε να ε, γίνουν οι εξή αλλαγέ μέσα σε διάταξη. Η δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το πολιτέ πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δημοκρατών Δικαιωμάτων για την περίοδο 2018-2022. Αυτό θα αντικατασταθεί ω θέμα από δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Πάντως ο τίτλο θα μείνει ο ίδιο, αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση. Οπότε τροποποιείται έτσι μέσα σε διάταξη η νομική επιτροπή ενέκρινε μια έκθεση για την κυρία Χάουτα, σύμφωνα με το άρθρο 9 8 του κανονισμού μας. Πρόκειται κατά τις ψηφοφορίες της Πέμπτης να ε, ψηφιστεί αυτό το κείμενο που αφορά την ασυλία της κυρίας Χάουτα. Επομένω και αυτή η αλλαγή στη μέση διάταξη εγκρίνεται.